υποβληθούν μέχρι την επόμενη περίοδο συνόδου. Θα αποστείλω τα όσα ψηφίσατε σήμερα στους αρμοδίους, διακόπτεται η περίοδο συνόδου και κλείνει η συνεδρίαση.